Colleagues, can I bring the meeting to order? Αρχίζουμε αγαπητοί συνάδελφοι. Να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη πρώτα απ' όλα, την έχετε μπροστά σας φαντάζομαι. Συμφωνείτε? Ανακοινώσεις. Πρώτον, στις 10 Φεβρουαρίου δεν θα συνεδριάσουμε. Θα συνεδριάσει όμως η Επιτροπή το πρωί μόνο της 11ης Φεβρουαρίου. Οι συντονιστές θα συνεδριάσουν τότε στις 10 του μηνός. Έτσι για να μην κάθονται, να δουλεύουν. Λοιπόν, στις 10 του μηνός μόνο συντονιστές. Το πρωί μόνο θα συνεδριάσει η Επιτροπή και μετά μόνο οι συντονιστές. Το άλλο για το οποίο θέλω να σας ενημερώσω, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι για το πακέτο που ο εισηγητής και ο σκιώδης εισηγητής ζήτησαν να ξαναδούμε τις τροπολογίες στις 17 Μαρτίου και η ψηφοφορία είναι στις 18 Μαρτίου. Οπότε 17 του μηνό θα εξετάσουμε τις τροπολογίες και θα ψηφίσουμε στις 18 Ψηφοφορίες τώρα. Έχετε τις κάρτες μαζί σας. Όχι βίζα, έτσι βάλετε τη βίζα, δεν δουλεύει στα μηχανήματα. Μόνο κάρτες ψηφοφορίες, οι οποίες ούτε και αυτές βέβαια δουλεύουν στα ATM. Για να κάνουμε μια δοκιμαστική ψηφοφορία πρώτα. Βάλτε τις κάρτες σας. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Ε, εντάξει. Μήπως υπάρχει κανείς που δεν έχει μαζί την ε, κάρτα του. Ντάβιτ, την έχεις, της έχεις. Ωραία. Όλοι. Έχετε τις κάρτες σας, εντάξει. Η κυρία Μάστρομ και ο κύριος Γκρός, τι λέτε, να συνεχίσουμε, μας αφήνετε, ωραία. Κάνουν διαπραγματεύσεις για το transfer. Μπορείτε να αγοράσετε έναν από την Τζέλση αν έχετε 38 εκατομμύρια να δώσετε. Ψηφίζουμε. Έτοιμοι. Συμβιβαστική τροπολογία 1. Υπέρ. Α, συγγνώμη, συγγνώμη. Προηγουμένω. Πρόκειται για την πρόταση Κανονισμό όσον αφορά την υλοποίηση του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού. Αναδιατύπωση, έτσι. Συμβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 145 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 146 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 147 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε. 147. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε. Πάλι το Γιβραλτάρ έχουμε μπροστά μας, φαίνεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα της φοφορίες. Εγκρίνεται περίεργα τα νούμερα. 148 και 142 υπέρ, κατά, αποχές, το ίδιο αποτέλεσμα. Εκατόν πενήντα τώρα. υπέρ, κατά, αποχές, θα ελέγξουμε. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι, πέρα στις ουφορίες. Εγκρίνεται. 151 και 153 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 152 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 19 υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ για την 19. Ψηφίσατε όλοι πέρα της ψηφοφορίας εγκρίνεται. 20 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 21 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 154 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 23 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 24 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 155 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 25 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 156 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 157 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 158 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 159 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 160 ως προστίκη υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 161 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 26 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 162 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 164 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 163 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 165 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. «187 τώρα» της κυρίας Φώστερ και «188 Παρνιό υπέρ» κατά αποχές απορρίπτονται. 47 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε για την 47. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι πέρα τη ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 48. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 49. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 189. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 190 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε. 189. 190 διορθώνει τώρα ο πρόεδρος. 190. Ηλεκτρονικά ψηφίζουμε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. 53 Πρέπει να αλλάξω τα γυαλιά μου, λέει ο πρόεδρος. 53 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 54 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 55 υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε. 55. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι πέρα τη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 191 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 56 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 192. Θέλετε να ελέγξουμε. 192 υπέρ, κατά, αποχές. Αυτήν θα την ελέγξουμε. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι πέρα της ψηφοφορίες. Εγκρίνεται. Νομίζω όντως εγκρίνεται. 57. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε. Νομίζω ότι απορρίφθηκε, αλλά θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. 57. Ψηφίστε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα στις ψηφοφορίες. Απορρίφθηκε. Με την ίδια πλειοψηφία. 58 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. 193 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 194 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 197 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 63 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 198 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Μαζί τώρα 67, 68, 69 και 70 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνονται. 201 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 202 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 5 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 74 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 205 ως προσθήκη υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 206 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 207 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 237 του κύριου Γκάλερ. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 239 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 241 καταπίπτει, 238 προσθήκη, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 240 επίσης προσθήκη, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 77 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 242 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 243 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 131 131 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 130 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 79 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 250 προσθήκη υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 248 και 249 μαζί είναι οι ίδιες προσθήκη υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. 80. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 251 και 252. Όχι. Καταπίπτουν. 254. Παρνιό τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 81. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 253 κατά πίπτη. 255. Παρνιό. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 258. Υπέρ. Κατά Αποχές απορρίπτεται. 257 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 256 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 260 γκάλερ υπέρ. Κατά. Αποχές Απορρίπτεται. 82 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 259. Καταπίπτει. 261 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 83 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 262 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 263 προσθήκη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 264 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 265 και 266 που είναι ίδιες υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 267 προσθήκη. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 86. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 268 και 269 που είναι ίδιες, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. 85, 87, 88, 94. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. 270 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 272 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε παρακαλώ για το 272. Ψηφίστε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. 271 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 273 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 274 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 275 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 277 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 276 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 278 υπέρ θέλετε να ελέγξουμε για τη 276. Ωραία, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για τη 276. Ψηφίσατε όλοι πέρα τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται με μία ψήφο διαφορά. 278. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 279 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 280 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 92 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 281 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 93 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. ...282 υπέρ... ...κατά... ...αποχές εγκρίνεται... ...283, 284, 285... ...μαζί... ...υπέρ... ...κατά... ...αποχές εγκρίνονται... 96 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 286 προσθήκη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 97 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 287 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 289 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 288 προστίκη υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 290-291 που είναι ίδιες μαζί υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. 292 καταπίπτει, 308 τώρα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 293 και 295 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται. 294 υπέρ, κατά, αποχές θα ελέγξουμε. 294 πάλι με μια ψήφο μάλλον θα είναι διαφορά. Ψηφίζουμε λοιπόν. Η ηλεκτρονικά ψηφίσατε όλοι, πέρα στις βοφορίας. Παραπάνω ήταν η διαφορά. Εγκρίθηκε. 296 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 297 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 99 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 298 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 299 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 300 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 301 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 302 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 303 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 304 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 100 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 101 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 305 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, αλλά ας ελέγξουμε καλύτερα. Ψηφίστε παρακαλώ για την 305. Πέρας της φοφορίας εγκρίνεται με μια ψήφο διαφορά. 306 υπέρ, κατά, 306 είπα, υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε για την 306. Ψηφίστε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι πέρα της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται με μια ψήφο δύο φορά. Φανταστείτε στην Ολομέλη θα 307 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 103 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 104, 1 και 5 μαζί υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται. 309 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 310 και 312 μαζί υπέρ, κατά, αποχές θα ελέγξουμε. 310 και 312, έτσι, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά, ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι πέρα τη υποφορία. Εγκρίνεται. 311 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 313 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 314 προσθήκη υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 315 υπέρ κατά, αποχές απορρίπτεται. 107 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 10 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δύο σελίδες ακόμα, 2, 20 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 321 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 323 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 324 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 325 υπέρ, κατά, αποχές, ηλεκτρονική επαλήθευση, άρτη ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι, πέρας. Απορρίπτεται. 109 υπέρ. κατά, αποχές, εγκρίνεται. 326 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 112 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 114 υπέρ, κατά, αποχές, ηλεκτρονική επαλήθευση για την 114 άρτη ψηφοφορία, Ψηφίσατε όλοι, πέρας. Ισοψηφία απορρίπτεται 115 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 116 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 117 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 118 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 3 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 121 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 11 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 127 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 4 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 129 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 132 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση για την 132 άρτη ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. 133 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 134 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 135 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 139 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 9, αποσύρεται, 10 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 140 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 141 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 143 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Κύριε Ρος, πριν τελική ψηφοφορία. Σύντομα, Πρόεδρε, στη συμβιβαστική υπαριθμών 8 θα έπρεπε να ψηφίσουμε από κοινού και τη συμβιβαστική 12. Εσείς όμως ε, ζητήσατε να ψηφίσουμε μόνο το συμβιβασμό 8 και όχι και τον 12. Άρα πρέπει να ψηφίσουμε ακόμα και τη συμβιβαστική 12. it's one vote, oui, mais il doit le dire, c'est le parce que c'est les No, you're absolutely right. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ήταν ταυτόσιμε συμβαστική 8 και συμβαστική 12, γι' αυτό προχώρησα κατά αυτόν τον τρόπο στην ψηφοφορία. Πάντω ψηφίζουμε τη συμβαστική 12 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Πολύ ωραία. Περνάμε στη τελική ψηφοφορία. Άρτε ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 26 υπέρ, μία ψήφος κατά και τέσσερις αποχές. Εγκρίνεται λοιπόν το νομοθετικό ψήφισμα υπέρ. Άρτη ψηφοφορία μάλλον. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 26 υπέρ, μία ψήφος κατά τέσσερις αποχές και εγκρίνεται. Συγχαρητήρια κύριε Μαρινέσκου. Περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Περνάμε στην ενημέρωση από τους τριμερείς διαλόγους, λέει ο Πρόεδρος. Συγγνώμη, συγγνώμη, λέει ο Πρόεδρος. Ξέχασα ότι έχουμε να ψηφίσουμε την έκθεση του κυρίου Σάσολη. Σας ζητώ συγγνώμη, λέει ο Πρόεδρος. Ναι, ναι, το βρήκα. Τώρα το βλέπω στη μερίσια διάταξη, λέει ο πρόεδρος. Περνάμε στην έκθεση για την τροποποίηση του κανονισμού 216, κάθετος 2008, όσον αφορά τα αεροδρόμια, τη διαχείριση της νέας κυκλοφορίας και τις υπηρεσίες αεροναυτιλίας. Η συγκητής είναι ο κύριος Σάσολη. Τροπολογία 29 και 30 μαζί. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. 31 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 32 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 8 και 9 μαζί υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση για τις τροπολογίες 8 και 9. Άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτονται. Περνάμε στην τροπολογία 38. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 39 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 40 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 41. Μάλλον 42 λέει ο πρόεδρος. Όχι, τη 41 ψηφίζουμε υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται. 42 υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται. 43 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. 44 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. 45 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 46 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 47 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 48 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 49. Δεν την ψηφίζουμε γιατί έχει, έχουμε καταψηφίσει τη 48 ούτε την 50, 51, 52, 53 δεν τις ψηφίζουμε, πάμε στην 54 υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται, 55 έχει αποσυρθεί, η 56 είναι τεχνικής φύσεως, περνάμε στις τροπολογίες 57 έως 64, όλες μαζί υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. Έχει αποσυρθεί η τροπολογία 65. μια προφορική τροπολογία από τον κύριο Σάσολη. Ο κύριος Σάσολη, κύριε Πρόεδρε, υπάρχει ένα πρόβλημα τεχνικής φύσεως. Στην τροπολογία 65 Ζητάμε να διαγραφούν τα National Aviation Authorities, η διατύπωση αυτή, στο άρθρο 1 σημείο 17F της πρότασης κανονισμού 216 του 2008 ζητάμε επίσης την παράγραφο 7 να γίνει μια αλλαγή όσον αφορά την δεύτερη υποπαράγραφο και να αντικατασταθεί διατύπωση από αυτό το οποίο ακολουθεί, is replaced by the following στην τροπολογία. Υπάρχει κάποια αντίρρηση για την προφορική αφιτροπολογία. Όχι υπέρ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 66. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 67. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 68 Η 38 είχε απορριφθεί, άρα δεν ψηφίζουμε την 68. 11 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 69 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 70 και 71 μαζί υπέρ, κατά, αποχές, ηλεκτρονική επαλήθευση και αυτές τις δύο τροπολογίες, 70 και 71, άρτη ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Είστε σίγουροι ότι ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτονται. 72-73 μαζί υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτονται. 74-76 μαζί υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτονται. 75 και 77 μαζί υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτονται. 78 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 79 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 80 και 82 μαζί υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 81 και 83 μαζί υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 85 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 14 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 15 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 2 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. «105» μάλλον συμβαστική τροπολογία 3 πρώτα, Συμβασική τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 3. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 105. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 19 υπέρ. Κατά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 κατά, αποχές, εγκρίνεται. 23 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 4 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 25 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 109 υπέρ, κατά, αποχές,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 Με την προφορική λοιπόν τροπολογία η 6 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία, άρτη ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι, πέρας. 29 υπέρ, μία ψήφος κατά, καμία αποχή, εγκρίνεται. Νομοθετικό ψήφισμα, άρτη ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 28 υπέρ, μία ψήφος κατά, καμία από εκεί. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια κύριε Σάσολη. Now we go into camera for the report on the Και κλεισμένο τώρα το θυρών, ενημέρωση για τους τριμερείς διαλόγους. Ζητώ συγγνώμη από τον κύριο Σάσολη, παραλίγο να μην ψηφίσουμε την έκθεσή του ένα μικρό λαθάκι δικό μου, λέει ο Πρόεδρος. Αποχωρήστε, παρακαλώ πολύ, από την αίθουσα όσοι δεν μπορείτε να μείνετε για τη συνεδρίαση και κλεισμένων των θυρών. Σας ευχαριστώ.